σε 20, 30, 50 χρόνια τα παιδιά μας ε, θα ζουν ακόμη και θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους προσφέρουμε ένα καλό, καλύτερο μέλλον και να διαφύγουμε από αυτό το κλίμα κρίσης στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ωραία, περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Θα έχουμε κάτι παραπάνω από μια ώρα. Παρακαλώ να συγκεντρωθείτε. Να συγκεντρωθείτε, εάν θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς, να μου το ζητάτε, αλλά με τη μέγιστη δυνατή συνεργασία. Σας αναγγέλω, όπως ε, υπόθηκε και αποφασίστηκε από την διάσκεψη των Πρόεδρων, σήμερα δεν προβλέπονται αιτιολογήσεις ψήφου προφορικές, διότι θα τις ακούσουμε αύριο. Έκθεση Αλφόνση. Ε, ονομαστική ψηφοφορία. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ο εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο πριν την ψηφοφορία. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Εάν θέλετε να προχωρήσουμε ήσυχα, θα πάρω όλα καλά. Αλλιώς θα χάσουμε δύο ώρες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Πολύ σύντομα, η γλωσσική πολυμορφία, το αντικείμενο αυτή τη έκθεση είναι ουσιαστική διάσταση τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση, κάτι που το επιβεβαιώνει και η συνθήκη τη Λισαβόνη, η οποία θέλει να ε, αναπτυχθούν και να ανθίσουν οι πολιτισμοί τη Ευρώπη σε περιφερειακό και ε, τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να αντιδράσει ε, ως προς την εξάλληψη πολλών δεκάδων γλωσσών που απειλεί την Ευρώπη, κάτι που επιβεβαιώνει ο στόχο και η UNESCO. Ε, είναι πραγματικά ένα μέρος του πολιτισμού της Ευρώπης που χάνεται όταν χάνεται και μια γλώσσα. Θα πρέπει η έκθεση λοιπόν να τονώσει τη δράση που να αναλαμβάνεται προ αυτή την κατεύθυνση. Και η σύνταξη της έκθεσης αυτής έγινε με τη συμμετοχή πολλών ομάδων, οπότε έτυχε και της ομόφωνης ψηφοφορίας της και από την Επιτροπή Πολιτισμού. Θα θα ήθελα λοιπόν να κλείσει με αυτόν τον αίσιο τρόπο και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στο το Κοινοβούλιο, να δώσει μια νέα δυναμική όθηση στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών γλωσσών που απασχολεί εκατομμύρια πολίτε στην Ευρώπη, προκειμένου να διατηρηθεί και ο πολιτισμό και η παράδοση των προγόνων του και να μπορέσουμε αυτόν τον πολιτισμό να μεταδώσουμε και στι πολιτικέ γενναίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Γκρότε. Υπέρ. Κατά. Ποιος απέχει. Εγκρίνεται. Έκθεση Λαβία. Ονομαστική άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη έκθεση Λαβία, δηλαδή, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λαβία Βον. Ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φερνάντε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λαβία. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα παρακαλώ να επιτείνετε την προσοχή σας, διότι θα έχουμε μια περιπλοκότατη ψηφοφορία. Έκθεση Λεπάζ. 50 τροπολογίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Παρακαλώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε. Να σας πω το Σε σχέση με τον κατάλογο ψηφοφορίας του ΕΛΚ στην τροπολογία 60 60 υπάρχουν υπάρχει μια χωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι ονομαστική ψηφοφορία ε, το έχουμε σημειώσει ως ε, ψηφοφορία κλειδί. Το δεύτερο μέρος που επίσης είναι ονομαστική ψηφοφορία επίσης θα έπρεπε να είναι ε, ψηφοφορία κλειδί. Ενώ δεν το έχουμε σημειώσει. αλλά θα έπρεπε επίσης να είναι. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 60. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ψηφίζουμε λοιπόν από κοινού 50 τροπολογίες. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 13 τροπολογίες της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ομαδική ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. απορρίπτονται. Επιτροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι σαφές ότι απορρίπτεται, αλλά αν θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Είναι σαφές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Ελέγχουμε για τη 44. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Έλεγχος για το 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα έλεγχος για το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Παρακαλώ όμω να υψώνετε τα χέρια σα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Έλεγχο. Παρακαλώ, έλεγχο. Να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Σας προκαλώ να είστε πιο συγκεκριμένοι. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά, έλεγχος παρακαλώ. 138 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Έλεγχο για το 140. Εντάξει λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Όντως απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. Με μία ψήφο διαφορά. 41 υπέρ. Συγγνώμη, 184 υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ να υψώνετε τα χέρια σας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 144 Ονομαστική ψηφοφορία. Μάλλον ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται, πέρας. «42 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. πέρας, απορρίπτεται». 60 σε τρία τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο μόνο τελικά. Αυτοδιορθώνομαι. 188 καταπέπτει. 147 έλεγχος, γιατί δεν, δεν τα χέρια σας, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. 63 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα της 63. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Αγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 ονομαστική ψηφοφορία, ε, άρχιτη ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε άρχιτη ψηφοφορία πέρας Απορρίπτεται. Τροπολογία 152 σε τρία τμήματα. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167 καταπίπτει. 167 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. 152 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 177 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 181. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 178. 178. Καταπίπτη 81. Καταπίπτει. 152. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 167 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. 185. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. 82 κατά καταπίπτει. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 187 μάλλον. 153 Έλεγχος για την 187. Άρχεται, πέρας. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86-87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, εγκρίνεται συγγνώμη 67 υπέρ κατά α, έλεγχος άρχεται η ψηφορία πέρας απορρίπτεται 169-171 με συγχωρείτε 140 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορείτε να υψώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Έρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 169-171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 172. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 157. Υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 107 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για το τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνατε. 190 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται. 179. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159. Άρχεται ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. 167. 161 ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112. 111 έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 112. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 113. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 114. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 115. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 116. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Καταπίπτει 162, 117. Μονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 118 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 119 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος για την 163. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 120. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 164 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 186. Προπολογία της εισηγητρίας. Παρακαλώ. Η συγκίτρια...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 Ευχαριστώ. Καταπληκτικά. Ευχαριστώ την τεχνολογία. Προτείνω μια προφορική τροπολογία. Σας προτείνω να εξαλείψουμε, να καταργήσουμε τη διαγραφή του μικρού β του ε, παραδείγματος 9 που αφορά τα υλικά κυταρίνης σε ότι ε, και αυτές οι εξαιρέσεις να συμπεριληφθούν στο α του 9. Είναι πολύ τεχνική παρατήρηση, ιδιαίτερος τεχνική αλλά ο στόχος είναι αυτά τα υλικά της κυταρίνης να συμπεριλαμβάνονται στα, στη λίστα των προηγμένων καυσίμων. Ελπίζω να είναι σαφές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, να ψηφίσουμε όπως το πρότεινε η συγκεκριά. 186 υπέρ. Κατά, αποχές, ξανά, υπέρ. Κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Εγκρίνεται. 180. Έχει αποσυρθεί. 121 και 167 καταπίπτουν τη σκέψη 1. Όχι, όχι. Ε, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6, όχι με συγχωρείτε. Τροπολογία 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Εκα... Ε, τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ Α, να ελέγξουμε. Ελέγχουν την 124. Άρχεται. Εγκρίνεται. Ε, εγκρίνεται. Τρεις ψήφοι. 7 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 127 κατά πίπτη, 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ. Α, θέλετε να ελέγξουμε τα 128. Πέρας. Απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος 130 πέρας απορρίφθηκε 175 καταπίπτει 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο? Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά Άποχες. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 183 έλεγχος άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Α, καταβήκεται κανένα. 134 υπέρ κατά αποχές. Α, έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 22 τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα πίπτη. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133-139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Α, έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται πέρας απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρας απορρίπτεται ισοψηφία 339 339 ψήφι Και τώρα η πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η εισηγήτρια θέλει να πάρει το λόγο εκ νέου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας προτείνω να αναβάλουμε την ψηφοφορία του νομοθετικού ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 57.2 του κανονισμού να μου δώσει την εντολή να διαπραγματευθώ. κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Ήταν πολύ επίμαχη έκθεση. Η ομάδα μου θέλει οπωσδήποτε να υπάρξει δεύτερη ανάγνωση. Γι' αυτό παρακαλώ να μην δεχθείτε αυτή την πρόταση. Ωραία. Ψηφίζουμε την πρόταση της εισηγήτριας. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Έλεγχος. Αν και θεωρώ ότι απορρίφθηκε. Άρχεται. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε μία ψήφος διαφορά. Quindi... Οπότε ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ονομαστική ψηφοφορία Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Λόβιν. Παρακαλώ λίγη στοιχεία για να προχωρήσουμε. Έξι τροπολογίες της Επιτροπής ΕΝΒΙ υπέρ. Παρακαλώ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Παρακαλώ, Παρακαλώ, ε, ησυχία. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Σα παρακαλώ ε, ε, να υψώνετε τα χέρια σα γιατί ε, θα καθίσουμε ακόμη περισσότερο. Τροπολογία 7 υπέρ κατά Αποχέ. Έλεγχο. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Α, ελέγχουμε την 9. Ωραία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία α καλά ελέγχουμε την 11 πέρας εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 Έχουμε εδώ προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να γίνει μια αλλαγή στην ε, ημερομηνία στο άρθρο αυτό. Αντί για 31 Οκτωβρίου, 31 Δεκεμβρίου 2013, μια που είναι ήδη Σεπτέμβρης, δεν προλαβαίνει η Κομισιόν να κάνει μια νέα αξιολόγηση. Δεν έχει κανείς αντίρρηση. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε, τη 14. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 16. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται να το επαληθεύσουμε την τροπολογία 19 πέρας της ενσφοφορίας απορρίπτεται τώρα έχουμε την πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και το Σχέδιο ψηφίσματο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Λεγκρίπ. Ε, μπλοκ 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το μπλοκ 2 καταπίπτει. Έχουμε λοιπόν μονομαστική ψηφοφορία την πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα με ονομαστική ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται έκθεση σκοτά μπλοκ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μπλοκ 2 καταπίπτει πρόταση της Κομισιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται έκθεση γκρότε Ο εισηγητής θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω, συνάδελφε, αλλά πριν πάμε να φάμε, πρέπει να, πριν πάμε στο μεσημεριανό, πρέπει να ψηφίσουμε τις πέντε οδηγίες του πρωινού. Αλλά το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος δηλαδή, περιμένει ακόμα την δημοσίευση των νομοθετικών κειμένων. Δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση. Ανεπισήμως μας έχουν πει πως θα γίνει κάτι τέτοιο εντός ενός μηνός. Αυτό κάποιοι συνάδελφοι δεν το θεωρούν σωστό. Οπότε θέλουμε να ψηφίσουμε μπλοκ 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, μπλοκ 2 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την πρόταση της ε, Κομισιόν. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Με ονομαστική ψηφοφορία το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Τσανώνη. Ο κύριος Χουντής ζητάει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ομάδα μου στη διάσκεψη των Προέδρων είχε προτείνει να μπει αυτό το θέμα και να πάμε για ψηφοφορία αφού συζητήσουμε. Σας λέω όπως ξέρετε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είμαι ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας το 85% των αναφορών έχουν σχέση με το ζήτημα που συζητάμε δηλαδή με τις δυσμενείς επιπτώσεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων η επιτροπή αναφορών δούλεψε με πάρα πολύ σοβαρότητα και θα ήθελε να ακουστεί η άποψή της δυστυχώς εισήχθη χωρίς τη σχετική συζήτηση. κατόπιν τούτου κυρία πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι προτείνω αν είναι να γίνει συζήτηση να ακούσουμε και τη γνώμη της επιτροπής και να μπορέσει και το κοινοβούλιο να τοποθετηθεί υπεύθυνα σε πολύ κρίσιμες ρυθμίσεις για τις οποίες ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ασκούνται πιέσεις προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση προτείνω το θέμα να συζητηθεί στην ολομέλεια του οκτωβρίου με συζήτηση και ψηφοφορία με την προϋπόθεση ότι θα γίνει συζήτηση ουσιαστική σας ανέφερα τους λόγους. ευχαριστώ κυρία πρόεδρε θέλετε να αναβληθεί για την πρώτη λομέλη του Οκτωβρίου. Χρειάζεται όμως ένας εισηγητής να είναι υπέρ. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις ή συμφωνία, αλλιώς ψηφίζουμε. Δεν βλέπω να υπάρχουν εδώ εισηγητές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Relazione Gabriel, per appello Έκθεση Γκάμπριελ. ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση Γκάμπριελ. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Παπα-Νικολάου. Παράγραφος 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 34. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Με ονομαστική ψηφοφορία μάλλον. Α, υπέρ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Παράγραφος 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 52, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 62. Υπέρ. Κατά Μάλλον ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία υπέρ. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 63 από το τμήμα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 67 δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρας άρχεται ε, εγκρίνεται συγγνώμη το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας Εγκρίνεται. Έκθεση στη Γκλεύσκα. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 16, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 19, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21, δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 25, πρώτο τμήμα, ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ,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 σε δύο τμήματα, σε τρία τμήματα μάλλον. Ε, πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται, πέρας, εγκρίνεται παράγραφος 44, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, Τροπολογία 1. Πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Έλεγχος. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Όχι. Παράγραφος 57. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος πέρας της προφορίας εγκρίνεται 58 τρία τμήματα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τρίτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 60, υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 67 σε τρία τμήματα. Υπέρ, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο, Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική μάλλον ψηφοφορία. Άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστική. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 68. Ε, Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. 74 από το τμήμα. Ε, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 76 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 82, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 84 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G. πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη S. Ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα το σύνολο της πρότασης, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Κοράτσα Μπίλτ. Χειροκροτήματα. Έκθεση Κοράτσα Μπίλτ. Τροπολογία 9. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Α, μα, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύρια Κοράτσα Μπίλτ. Εκτός μικροφώνου. Πολύ σύντομα σας ευχαριστώ. Θέλω να απευθύνω έκκληση στους ε, συναδελφούς να ψηφίσουν υπεύθυνα υπέρ της οδηγίας αυτής ε, των υπηρεσιών. Ε, να το καταψηφίσουν σημαίνει ότι θα καταψηφίσουν τις θέσει εργασία στην Ευρώπη. Λάβουμε υπόψη όλες τι ανησυχίες των ε, σοσιαλδημοκρατών για την κοινωνική διάσταση. Τα έχουμε καλύψει όλα ε, ό,τι αναφέρει η συνθήκη και η οδηγία υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Allora, possiamo procedere al voto. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 9, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Η ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 ονομαστική, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρα. Απορρίπτεται. 8. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελευταία έκθεση. Παρακαλώ την εισηγήτρια. Πρόεδρε. Η πράσινη δυστυχώς και άλλες ομάδες καταψήφισαν αυτή την έκθεση και αυτό είναι ανεύθυνο. Ωραία. Προχωρούμε στην επόμενη έκθεση. Κυρία Γκέπχαρτ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ως σοσιαλδημοκράτες δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε έκθεση στην οποία ακυρώνεται η κοινωνική διάσταση των υπηρεσιών. Απορρίπτω αυτά τα οποία είπε η κυρία Κόρατσαμπιλτ. Ωραιότατα. Μενέντες Δελβάλε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος θέλετε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Το σύνολο του ψηφίσματος, όπως το αποποιήθηκε υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ για την άρεστη συνεργασία. Διακόπτεται η συνεδρίαση έως τις 2.30.